για τόσο σημαντικές ε, συναντήσεις ε, στο Συμβούλιο, βεβαίως και θα έπρεπε προηγουμένως ο κύριος Βαν Ρομπόε να έρχεται εδώ στο Κοινοβούλιο. Εντάξει, θα ενημερώσω για την ε, άποψη του Κοινοβουλίου και βεβαίως θα προσπαθήσω να είμαστε παρόντες και στην τελική φωτογραφία. Λοιπόν, όσον αφορά την ημερήσια διάταξη δεν υπάρχουν αλλαγές, γι' αυτό και θα περάσουμε στο πρώτο σημείο της ε, ημερήσια διάταξη. έκθεση Μπουζουτήλ. Πρόκειται για τον πίνακα... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόσφατα είναι μεγάλη κουβέντα για την ε, ανάπτυξη και το πώ θα δώσουμε κάποια όθηση στι οικονομίε τη Ευρώπη, ώστε να μπορέσουν να βγουν από αυτό το σημερινό διέξοδο. Όμω θα πρέπει να πάμε πέρα από αυτά τα συγκεκριμένα και θα πρέπει να πούμε με πιο συγκεκριμένο τρόπο το πώ θα επιτύχουμε αυτή την ανάπτυξη. Στη έκθεση μου αφορά τον πίνακα επιδόσεων αυτή τη ιστορική αγορά. Αυτό σήμερα και θα θέλω να σας πω ε, ένα σημαντικό μήνυμα, ότι αν θέλουμε να πετύχουμε την ανάπτυξη θα πρέπει τότε να μπορέσουμε να φέρουμε πιο κοντά την ενιαία αγορά ή στους πολίτες, γιατί είναι η πιο ε, σημαντική επένδυση της Ευρώπης για την ανάπτυξη. Οπότε θα πρέπει να επισκευάσουμε, θα πρέπει να, να, να ότι δεν δουλεύει καλά και, και να δούμε που δεν πετύχαμε. Κοιτάξτε, αυτός ο πίνακας αποτελεσμάτων μας δείχνει ότι μία σειρά των μελών ε, καταβάλουν κάποιες... Ε, ε, προσπάθειες για να μεταφέρουν. Κύριε Μπουζούτιλ διακόπτει ο Πρόεδρος. Κύριε ναι, ναι. περιμένετε παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, για όλους όσους δεν θέλουν να ακούσουν τον κύριο Μπουζουτήλ θα ήταν ίσως ε, ε, ευγενικό να εγκαταλείψετε την αίθουσα αυτή με ησυχία. Μπουζουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκείνου που προτίθενται να με ακούσουν τώρα. Μόνο εάν τα κρατη θέλουν να αναβαθμίζουν προσπαθία του ώστε να εξασφαλίσουν ότι γίνεται ορθή μεταφορά στο εργοδίκαιο των ε, ε, κοινοτικών μέτρων, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε μια εσωτερική αγορά. Βέβαια, δεν είναι όλα μαύρα και άραχλα, διότι κάποια κράτη-μέλη έχουν δείξει μια συνεπή προσπάθεια όσον αφορά τι καλύτερε επιδόσει στην εσωτερική αγορά και η Μάλτα, η πατρίδα μου, για άλλη μια φορά έχει τι καλύτερε επιδόσεις όσον αφορά τη μεταφορά των περισσότερων ευρωπαϊκών νομοθετημάτων εγκαίρω. Έχουν τώρα και άλλα κρατημέλη όπω η Εστονία, τα οποία έχουν ε, πάρα πολύ θετικέ επιδόσεις για όλα τα θέματα ε, τέτοιου ε, πίνακα τέτοιου ελέγχου επιδόσεων τη εσωτερική αγορά. Οπότε τώρα το θέμα δεν είναι ότι αν έχει τον κανόνα. Το θέμα είναι ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, ο καθένα ε, και τα άλλα κρατούν εκτό από αυτά μπορούν να τα πάνε καλά. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώ θα γίνει η ορθή εφαρμογή, η ορθή ε, μεταφορά στο ιστορικό όσο γίνεται πιο έγκαιρα. Μόνο έτσι θα μπορέσουν οι πολίτε μα και οι επιχειρήσει μα να ωφεληθούν από την εσωτερική αγορά. Τα κράτη-μέλη επομένω αυτό οποίο χρειάζονται είναι πιο φιλόδοξου στόχου. Θα πρέπει επίση να τηρήσουν τι δεσμεύσει του. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλευρά τη θα πρέπει να συνεχίσει να είναι η εκτελεστική εξουσία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επομένω καλύτερα, γρηγορότερα να ασκεί την διαδικασία επί παραβάση όποτε χρειάζεται. Και γι' αυτό έχουμε και μια τροπολογία. Με τροπολογία αυτή διατυπώνουμε μια ιδέα για μια ε, γρήγορη συνοπτική διαδικασία ε, επί παραβάση και είναι δυνατόν και αυτόν τον τρόπο κανείς μπορεί να ενεργεί για αυτόν τον τρόπο όποτε χρειάζεται και αυτό να γίνει με τρόπο αμερόληπτο, με τρόπο μακριά από οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση. Τώρα, πέραν ε, του ρυθμιστικού πλαισίου, θα πρέπει να δούμε ότι δεν είναι αυτό ο μόνο τρόπο να έρθει πιο κοντά στο διαγράμμα του πολίτε. Γι' αυτό τώρα σα λέω ότι η έκθεση μου επίση επικεντρώνεται και στο πώ η ιστορική αγορά ε, με πιο άμεσο τρόπο θα αγγίζει επιχειρήσει και Ευρωπαίου. Και εν προκειμένου έχουμε εδώ το συγκεκριμένο ε, δίκτυο των μέσων πολιτικής λογικής επιτροπής το Solvit και, άλλα, και, και, τα άλλα μέσα πολιτικής που έχει η Κομισιόν να χρησιμοποιηθούν το ώστε να οδηγηθούμε σε αξιοποίηση αυτών των υπηρεσιών γιατί ακόμα υπάρχει αυτό, αυτό το απρόσωπο δίκτυο και πλέγμα υπηρεσιών που θα πρέπει να καταφύγουν οι πολίτε όταν έχουν κάτι να καταγγείλουν, κάτι για το οποίο να παραπονεθούν. Και οπότε θα πρέπει ομένω κάθε φορά ε, αντί να λύνουν το πρόβλημα που έχουν, να λύσουν το πρόβλημα το διαδικαστικό. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με ε, αυτές τις υπηρεσίες, να δούμε το, το ότι ε, αυτή η διαδικτυακή πύλη η Ευρώπη σας να είναι το κλειδί στην επιτυχία του εγχειρήματος τώρα αλλά θα πρέπει επίσης να δούμε και τι γίνεται όσον αφορά το προσωπικό το αντίστοιχο να έχουμε επομένως ε, αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλε τι ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε που να επεξεργάζονται τι καταγγελίε των Ευρωπαίων. Γιατί πρόσφατα ζητήσαμε πάρα πολλέ θυσίε από του Ευρωπαίου. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε το, την επιβίωση των οικονομιών μέσα από την κρίση. Έχουμε όμω την εσωτερική αγορά που είναι ο καλύτερο τρόπο τόσο να πετύχουμε την ε, ευημερία και την ανάπτυξη. Αυτά δηλαδή που προσδοκούν από εμά οι Ευρωπαίοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπούσου Τελειοπρόεδρος και τώρα. Κύριε Μπαρνία, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω όλους. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σιμών Μπουσούτιλ για μια τεράστια προσπάθεια την οποία έκανε με την στήριξη και την κατανόηση <clears throat> όλων των μελών της Επιτροπής ΣΥΝΚΟ Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και ιδιαίτερα τους συντονιστές. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε μια κρίση, σοβαρή κρίση. Χρηματοπιστωτική που δεν έχει τελειώσει, οικονομική που έχει και κοινωνικές συνέπειες. Βλέπουμε το πώς εξελίσσεται η κρίση αυτή. Πολλοί πολίτες θίγονται από την ανεργία, υποφέρουν. Πολλοί έχουν εξοργιστεί και εκφράζουν την οργή τους και η εσωτερική αγορά στην οποία αναφερόμαστε με την έκθεση του κυρίου Μπουσούτιλ στην ουσία βρίσκεται σε μια παράδοξη θέση θα έλεγα. Θα μπορούσε αν δεν προσέξουμε να είναι το πρώτο θύμα αυτού, αυτής της έκφρασης οργής μιας εθνικιστικής αν θέλετε αντίληψης προστατευτισμού ενώ ταυτόχρονα η εσωτερική αγορά είναι το βασικό ατού το οποίο έχουμε, το βασικό χαρτί που έχουμε για να βγούμε από την κρίση. Αυτό έχουμε προσπαθήσει να πετύχουμε και από την έκθεση Μόντι και μετά με την έκθεση Γκρέσ, με τη στήριξη του Κοινοβουλίου προσπαθούμε έχουν γίνει άνω των 50 προτάσεων, θα γίνουν τουλάχιστον άλλες 10 επιπλέον για να επανεκκινήσει η αγορά και όλα αυτά θα πρέπει να συνοδεύσουν θα έλεγα τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάκαμψη την οποία συζητούν αυτή την εβδομάδα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Σωστή διαχείριση των δημοσιονομικών από τη μία, ανάπτυξη από την άλλη με την εσωτερική αγορά, στοιχεία κάλλιστα σύμβατα και τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν από κοινού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χαίρομαι που ο κύριος Μπουσούτιλ υπογράμμισε ότι η εσωτερική αγορά είναι μια δεξαμενή ανάπτυξη. Αν πάνε καλύτερα τα πράγματα στην εσωτερική αγορά, κινητικότητα εργαζομένων, υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, επενδύσεις, ε, θα έλεγα ότι θα μας βοηθήσουν και θα μας δώσουν 3-4 βαθμούς ανάπτυξης επιπλέον για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα οικονομικά αυτός ο χώρος των 500 εκατομμυρίων πολιτών και καταναλωτών και 22 εκατομμυρίων μικρών κυρίως και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Πρέπει οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν τα μέσα τα οποία απαιτείται ε, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με το Solvit, με την ε, ιστοσελίδα και την πύλη ε, την αντίστοιχη ακριβώς για να βοηθήσουμε και τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες και τους ε, Ευρωπαίους καταναλωτές. Ο πίνακας επιδόσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάμε, το λεγόμενο scoreboard. Αυτός ο πίνακας τον οποίο θα προτείνουμε δύο φορές κατέτος από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας δείχνει σε κάθε κράτος μέλος το επίπεδο εφαρμογής της νομοθεσίας της ε, εσωτερικής αγοράς. Εδώ έχουμε περίεργα ποσοστά θα έλεγα ή μάλλον ενδεικτικά ποσοστά τα οποία οδηγούν και πρέπει να ε, οδηγήσουν τα κράτη-μέλη σε περαιτέρω προσπάθειες. Αυτός ο πίνακας επιδόσεων δεν είναι φυσικά το μοναδικό μέσο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι η μοναδική χορδή την οποία είμαστε έτοιμοι να σημάνουμε. Όχι. Η κρίση αυτή στην οποία προαναφέρθηκα μας έχει οδηγήσει στο να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα από κάποιες δυσλειτουργίες στα κράτη-μέλη μας και να εγκρίνουμε κάποιες νέες προσπάθειες και νέα μέσα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εν πλήρη διαφανεία και σε στενή συνεργασία και με εσά, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά με τα κράτη-μέλη για να δείχνουμε σε αιτήσια βάση τον απολογισμό της διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς με τελευταία έκθεση την ανακοίνωσή μας της 24ης Φεβρουαρίου. Στην επόμενη συνάντηση, συνεδρίαση του, Συμβουλίου Υπουργών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγγνώμη, τον μήνα Ιούνιο θα έχουμε την επόμενη έκθεση προσπαθώντας να ενισχύσουμε τη σωστή εφαρμογή της νομοθετικής αρχιτεκτονικής της εσωτερικής αγοράς. Δύο βασικοί άξονες θα χαρακτηρίζουν την ανακοίνωσή μας η ανάπτυξη. Δεν μπορούμε εμείς να διατυπώσουμε νέους κανόνες χωρίς να ασχοληθούμε βέβαια με τη σωστή τους εφαρμογή. Η νομοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται δεν είναι μόνο άχρηστη, αλλά πολύ συχνά είναι αντιπαραγωγική, δημιουργεί ελλείψεις ισορροπίας στις σχέσεις δύο χωρών, μια χώρας με τους γείτονες της, οι οποίες μπορεί να εφαρμόζουν με πιο σωστό τρόπο τα μέσα και τις δυνατότητες και έτσι να περιορίζονται οι δυνατότητες των πολιτών και των επιχειρήσεων μια συγκεκριμένης χώρας. Γι' αυτό ακριβώς προτείναμε εμείς να μειώσουμε το ανεκτό έλλειμμα από το 1% σε 0,5% στον τομέα της μη εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων και χαίρομαι που συμφωνεί ο κύριος Μπουσούτιλ. Δεν μπορούμε να ικανοποιηθούμε με ένα έλλειμμα μεταφοράς 1,2% και μάλιστα σε ορισμένες χώρες βρίσκεται το έλλειμμα αυτό σε 1,7%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασίες με τα κρατημέλη για να βελτιώσει και να εξορθολογήσει τη λογική της εφαρμογής ε, των νομοθετικών ρυθμίσεων της εσωτερικής αγοράς. Όπως είχα ανακοινώσει πήγα σε όλες τις πρωτεύουσες και συναντήθηκα με όλους τους ανωτάτους δημοσίους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για την <clears throat> οδηγία, τη μεταφορά στην χώρα τους, την οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες, για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είχα μια άμεση επαφή μαζί τους με τους ανώτατους αυτούς διοικητικούς υπαλλήλους φτιάξαμε μια task force με 500 υπαλλήλους για να συνεργαστούμε εν πλήρη εμπιστοσύνη και πιο αποτελεσματικά και μάλιστα θα συνεχίσω τις προσπάθειες αυτές και με τους εκπροσώπους των περιφερειών, γιατί σε πολλές από τις περιφέρειες, σε επίπεδο της πραγματικής οικονομίας, των τοπικών περιφερειακών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικάτων, υπάρχουν εξαιρετικοί, θα έλεγα, εταίροι και θα αναφερθώ στον επόμενο γύρο αυτό, τον οποίο θα κάνω στην ανακοίνωσή μας τον μήνα Ιούνιο. Τέλος, <clears throat> πιστεύω ότι αυτά τα μέσα αρρωγής και πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά θα πρέπει να είναι πραγματικά στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Έχουμε ορισμένα μέσα για μεγαλύτερη διαφάνεια, για μεγαλύτερη καθαρότητα, αλλά τα μέσα αυτά, αν θέλετε, έχουν αναπτυχθεί ελαφρώς άτακτα. Θα πρέπει λοιπόν τα πράγματα να ταξινομηθούν σωστότερα, να γίνουν τα μέσα πιο αποτελεσματικά η ιστιακή θύρα, η Ευρώπη σας ανήκει, θα συνεχίσει να λειτουργεί και θα βελτιωθεί. Ελπίζω επίσης ότι το Solvit, το οποίο είναι επαναστατικό ε, online σύστημα επίλυσης προβλημάτων με τις εθνικές διοικήσεις, θα λειτουργήσει καλύτερα σε όλες τις χώρες μέλη. Αυτά κυρίες και κύριοι, θα εορτάσουμε την 20, τα 20 γενέθλια της εσωτερικής αγοράς. Ε, δεν θα πρέπει σε αυτή τη φάση κυρίως τα γενέθλια αυτά να είναι νοσταλγικά ή μελαγχολικά αλλά αισιόδοξα και δυναμικά γιατί οι πολίτες περιμένουν ε, συγκεκριμένα ωφέλη για την καθημερινότητά τους. Αυτό είναι και το πνεύμα για αυτή τη συμφωνία για τη σωστή διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς. Ο καθένας στο δικό του ρόλο, οι κυβέρνηση το Συμβούλιο, η Επιτροπή, τα Κοινοβούλια, θα κάνουν θα έλεγα αυτά τα 20 γενέθλια της εσωτερικής αγοράς μια νέα στιγμή όθησης, μια νέα στιγμή δυναμικής για την ενιαία αυτή αγορά. Ελπίζω να το συζητήσουμε το θέμα αυτό ακόμα περισσότερο, όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά με τους εκπροσώπους και εταίρους της χώρες ε, μέλη αυτό θα είναι και το πνεύμα αυτή της εβδομάδας της ενιαίας αγοράς στα πλαίσια του φόρουμ της Κρακοβίας που είχαμε κάνει στο παρελθόν από τις 12 μέχρι τις 17 Οκτωβρίου και στο Κοινοβούλιο θα εορτάσουμε τα 20 γενέθλια θα συζητήσουμε το τι πάει καλά, το τι δεν πάει καλά στις περισσότερες χώρες, πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, να υπεπιδίσουμε την πολυδιάσπαση που χαρακτηρίζει μερικές φορές την κατάσταση, πώς θα προωθήσουμε το λεγόμενο Single Market Act καλύτερα και πώς θα εφαρμόσουμε τις πολλά υποσχόμενες νέες πρωτοβουλίες. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω την επικοινωνία μαζί σας γιατί αυτό θέλουν οι πολίτες, αυτό είναι το αίτημα των πολιτών με όλους τους κινδύνους προστατευτισμού και αναδίπλωσης εθνικιστικής είναι να ξαναβρούμε την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε τώρα με τους ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Σβάμπ, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε εδώ ότι η αγορά, η εσωτερική αγορά, όπως είπε ο Επίτροπος, δεν θα πρέπει να είναι το πρώτο θύμα της κρίσης, αλλά αντίθετα 20 χρόνια μετά την ίδρυση αυτής της ενιαίας εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν έτσι ώστε να ακολουθηθούν ενιαίοι κανόνες οι οποίοι θα μας οδηγήσουν σε επιτυχή αποτελέσματα. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Μπουζουτήλ ιδιαίτερα για την εργασία του γιατί πραγματικά η ετήσια έκθαση το του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να μας δείχνει ακριβώς πού βρίσκεται αυτή η εσωτερική αγορά. Αλλά 20 χρόνια μετά το ξεκίνημα αυτού του εγχειρήματο θα πρέπει πέρα από τις τελετές και τον εορτασμό που θα γίνουν στο τέλος του χρόνου αυτού να δούμε τι ακριβώς συνέβη αυτές τις 20 χρονιές και τι ακριβώς πρέπει να βελτιωθεί. Η έκθεση του συναδέλφου Μπουζουτήλ μας δείχνει ακριβώς ποια συνεχίζουν να είναι προβληματικά σημεία αυτού του εγχειρήματο. Έλλειψη διαφάνειας. Υπάρχει νομοθεσία, η νομοθεσία η οποία ενδεχομένως δεν μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, είτε μεταφέρεται με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχουν αριθμοί που δείχνουν πραγματικά αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα Υπάρχουν όμως αριθμοί οι οποίοι κρύβουν το κατά πόσο αυτό το κοινοτικό και κεκτημένο δεν ε, αντικατοπτρίζεται με σωστό τρόπο. Διότι ναι μεν έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, δεν εφαρμόζεται όμως με σωστό τρόπο. Επίσης, οι διαδικασίες ε, επιπαραβάσει. Γνωρίζουμε σήμερα ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τις διαδικασίες αυτές. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη είτε δεν μεταφέρουν τις οδηγίες, είτε δεν είναι σε θέση να τις μεταφέρουν ορθά, με σωστό τρόπο. Η αποτελεσματικότητα είναι πάρα πολύ ελλειπής. Ο ε, κύριος Μπουζουτήλ προτείνει λοιπόν μια κατηγορία διαδικασιών fast track με μεγάλη ταχύτητα έτσι ώστε αυτά τα συνεχιζόμενα προβλήματα και ελλείψεις να ξεπεραστούν. Η Επιτροπή θα πρέπει λοιπόν να μπορεί να έχει ένα σύστημα εποπτείας, παρακολούθησης ελέγχου των οδηγιών που έχουν ήδη μεταφερθεί από τα κράτη-μέλη, τα οποία όμως μεταφέρουν με λανθασμένο και λυπή τρόπο αυτή την νομοθεσία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να δούμε το κεκτημένο πώς έχει εφαρμοστεί. Θέλουμε πίνακε αντιστοιχία, θέλουμε συγκρίσιμα στοιχεία από το 2004 παραδείγματο χάρη να μπορέσουμε να συγκρίνουμε το τι έχει γίνει πραγματικά. Γιατί σήμερα βλέπουμε ότι χρηματοδοτούμε αυτή την δράση και δεν έχουμε συγκρίσιμα και σωστά αποτελέσματα. Και θα πρέπει αυτό να το διαλευκάνουμε. Των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κορέιαντε Κάμπος, για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, κύριε Αγαπητέ κύριε Επίτροπη Μπαρνιέ, οφείλουμε συγχαρητήρια προς τον κύριο Μπουσούτιλ για το έργο το οποίο επετέλεσε και για να μπορέσουμε να έχουμε εύρυθμη λειτουργία τη αγοράς αγορά, θέλουμε καλύτερε επιδόσει ανάπτυξη και οι καταναλωτέ ξέρουν, μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται όσον αφορά την αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχονται Οπότε έτσι θα προσαρμοστούμε στι απαιτήσει τη παγκοσμιοποίηση. Επομένω, ο ρόλο τη Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό όχι μόνο στη φάση την νομοθετική που θα πρέπει να είναι επαρκή, θα πρέπει να είναι δόκιμη, αλλά θα πρέπει κατά τον ίδιο τρόπο να μπορέσουμε να φροντίσουμε και το θέμα τη μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο. Και εδώ έχουμε τα προβλήματα συνήθω, διότι ενίοτε τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι η φάση τη μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο δεν πειράζει να γίνει μέσα σε δύο χρόνια. Όμω έτσι παραβλάπτεται η λειτουργία αυτή τη αγορά των ε, ε, τόσων εκατομμύριων Ευρωπαίων. Γιατί θα πρέπει επομένω να δούμε πώ θα λειτουργήσει κάθε η ευρωπαϊκή αγορά. Δεν θα πρέπει να γίνεται ανεπαρκή, δεν πρέπει να γίνεται λανθασμένη μεταφορά των ε, οδηγιών στο ιστορικό δίκαιο, γιατί έτσι έχουμε θέματα παρερμηνία, προβλήματα εφαρμογή. Επίση, αυτή η ανακοίνωση του 2011 όσον αφορά την διακυβέρνηση, ε, μέσα σε ένα έγγραφο κατά κάποιο τρόπο κωδικοποιεί αυτό το, το, το πώ θα πρέπει να γίνεται η διακυβέρνηση, η διαχείριση τη αγορά και έχουμε επομένω τώρα να έχουμε μια οπτική, μια αντίληψη πιο ολοκληρωμένη για την ε, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και ε, οι ιστορικές επιμέρους αγορές θα πρέπει να ελέγχονται, να υποπτεύονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, αυτό το δίκτυο Solvit θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ σε σχέση με κάποια νομική φύσεω μέτρα, ούτω ώστε έτσι να έχουμε καλύτερη λειτουργία τη εσωτερικής αγορά. Θα πρέπει να έχουμε μια κατάλληλη νομική βάση και έτσι το Solvit να το εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο, να μπορέσουμε έτσι να ανταποκριθούμε στις ε, προκλήσεις που υπάρχουν και επίσης να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύτερα την διαδικασία παραβάση και να δούμε ε, τι θα γίνει με αυτό το φόρουμ της ενιαίας εμιτόπισης της αγοράς που όπως πατήθηκε από τον συνάδελφο το 2012 συζητήθηκε αυτό στην Κρακοβία και αυτό το φόρουμ ιστορικής αγοράς, αυτό το οποίο μας το είπε και ο κύριος Μπαρνιέ, αυτή η εβδομάδα ε, τη ε, εσωτερική αγορά, θα είναι πάρα πολύ σημαντική ούτω ώστε να κάνουμε βήματα προ τα εμπρό για να άρουμε του φραγμού που υπάρχουν στην ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά, διότι πέραν των προβλημάτων των άλλων ε, θα μπορούσαμε να λύσουμε το εξή. Θα έχουμε στον ίδιο χώρο του νομοθέτε, του επιχειρηματίες, του καταναλωτέ. οπότε κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε ο καθένα να βάλει το λιθαράκι του στον προβληματισμό αυτόν του που τι πάει στραβά στην εσωτερική αγορά, πώς θα προοδεύσουμε, πώς θα κάνουμε βήματα προόδου. Οπότε με αυτή την ευκαιρία θα πρέπει να δούμε αυτή την ε, πρόταση του εισηγητή. Την διατύπωσε λίγο πριν γίνει η ψηφοφορία, πριν τελειώσει η διαδρομή η εξάμηνη, όσον αφορά το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε πιο αποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας επιφαραβάσεως. θα πρόκειται για κάποιον ο οποίος κάποιο τρόπο θα επιμελείται τις εσωτερική αγορές. Βέβαια θα πρέπει να εμβαθύνουμε τον προβληματισμό πάνω ε, σε αυτή την ιδέα. Να δούμε ποιο όργανο, ποιος θα αναλάβει αυτή την ε, αρμοδιότητα. Δυστυχώς η πρόταση αυτή κατέβηκε όπως είπαμε την τελευταία στιγμή κάποιο τρόπο όταν, όταν ολοκληρώνονταν η διαδρομή της ε, έκθεσης Οπότε θα πρέπει να δούμε πώ θα βρεθεί κατά πιο καταστήμα θα συζητήσουμε όλα αυτά. Ομάδα των Φιλελευθέρων, τον κύριο Γιώργο Χατζημαρκάκη, να πάρει το λόγο για 5,5 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κύριε Σιγητά, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα πραγματικά να χαιρετήσω την πρωτοβουλία του συναδέλφου, του κυρίου Μπουζουτήλ. Πρόκειται για μια πραγματική δυνατότητα που έχει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφραστεί και να πάρει θέση για τόσο σοβαρά θέματα. Πρόκειται για ένα πολύ επίκαιρο θέμα, καθότι η μεταφορά ορισμένων αρχών που οδήγησαν στην ίδρυση πριν από 20 χρόνια στην εσωτερική αγορά έχουν οδηγήσει σε κάποιες ανισορροπίες. Μπορεί κανείς να πει ότι σαφώς και κάποια από αυτά τα οποία δεν εφαρμόστηκαν σωστά έχουν μια βαρύτητα σήμερα στην οικονομική κρίση και κινδυνεύουμε να χάσουμε την αξιοπιστία μας, την νομιμότητά μας γιορτάζοντας ε, την 20η επέτειο της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει λοιπόν σήμερα να επιστήσουμε ιδιαίτερα τις ε, προσπάθειές μας και την προσοχή μας σε αυτές τις αδυναμίες που συνεχίζουν να υπάρχουν. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η εσωτερική αγορά βεβαίως και είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Κάθε χρόνο αποφασίστηκε να δημοσιεύονται οι αιτήσει εκθέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο στην εσωτερική αγορά. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι βεβαίως αυτοί οι οποίοι εγκαίρως και νωρίς μεταφέρουν τις κοινοτικές οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο να μην ε, τιμωρούνται. Σε καμία περίπτωση. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι επιτέλους στην ε, εσωτερική αγορά να μεταφέρονται όλες οι συγκεκριμένες οδηγίες μέσα στα χρονικά πλαίσια. Η ταχύτητα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική για την μεταφορά. Και βλέπουμε ότι από 5,5 μήνες που χρειαζόταν για την μεταφορά ενός νομοθετικού κειμένου στο Εθνικό Δίκαιο, έχουμε περάσει το 2011 στους 8 μήνες. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη και οι εθνικές αρχές να δεσμευθούν έτσι ώστε εγκαίρως να μεταφέρονται τα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα. Μετά από 20 χρόνια εσωτερικής αγοράς βλέπουμε ότι οι επιτυχίες όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειωθεί. Η ανταγωνιστικότητα αυτή έχει σημαντικά υποχωρήσει και η κατάσταση είναι δραματικά υπέρ των πιο ισχυρών. Βλέπουμε ότι η Επιτροπή των Χαμηλών Επιτυχίων έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλες ανισότητες, οι οποίες διαρκώς αυξάνονται. Εμείς σαν Ευρωπαίοι βρισκόμαστε στην καρδιά αυτού της προσπάθειας. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά να κοιτάξουμε αυτήν την ανταγωνιστικότητα η οποία δυστυχώς δεν βελτιώθηκε με αυτήν την οικονομική πολιτική. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά αυτός ο πίνακας αποτελεσμάτων αποτελεί μια ευκαιρία να βελτιωθεί η κατάσταση. Η 20η από την ίδρυση της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να γίνει ένας απολογισμός και σε εθνικό επίπεδο αλλά και ενδεχομένως σε μια περαιτέρω αποκέντρωση στις περιφέρειες. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε ίσως να αποκαταστήσουμε τις ανισορροπίες. Ο Νότος, ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση και υποφέρει από αυτήν την πολιτική. Κάνω λοιπόν μια έκκληση προς την Ευρώπη. Χρειάζονται νέες θεωρίες, νέες θεωρίες οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε περισσότερο ισορροπημένη ανάπτυξη και όχι σε μια αντιπαράθεση όπου οι ισχυροί διαρκώς δυναμώνουν. Πιστεύω ότι αυτή η 20η επέτειος της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε εμείς οι Ευρωπαίοι όλοι, όχι μόνο οι δυνατοί του Βορρά, να αντιμετωπίσουν με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον. Η Σιάρη θέλω να παρακαλέσω την κυρία Τζούλη Γκέρλινγκ να πάρει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Madam President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική μα ομάδα θέλει πάρα πολύ θετική την προσπάθεια αυτή τη έκθεση, γιατί όπως ξέρετε δεν σημαίνει αυτό πάντοτε από πλευρά μα, αλλά όμω πρόκειται εν προκειμένου για θέμα τη ουσιακή αγορά όπου όντω ε, χρειάζεται ε, να ενεργήσουμε με κάποιον ενθουσιασμό και με θετικές προσπάθειες να βοηθήσουμε να ολοκληρωθεί η ιστορική αγορά διότι και οι επιχειρήσεις όπως και οι καταναλωτές είναι αυτοί οι οποίοι θα ωφεληθούν από μια εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και το σούτο μάλλον ε, σε μια συγκυρία ε, δύσκολη όπως ε, σήμερα. Τι κάνουμε τώρα, κοιτάμε πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης να δούμε τι ευκαιρίες υπάρχουν για εξαγωγές, οπότε εν αυτή περιπτώσει δεν θα πρέπει να αγνοούμε και τις ευκαιρίες που παρέχονται εντός των σύνορων μας. Βεβαίω, το να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια τέτοια ιστορία για επιχειρήσει και για καταναλωτέ δεν είναι κάτι το οποίο απαιτεί μόνο ορθή εύστοχη νομοθεσία, χρειάζεται και σωστή συνέργεια, σωστή εφαρμογή από πλευρά των ε, κυβερνήσεων. Διότι χωρί να υπάρχει ορθή εφαρμογή, οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να ωφεληθούν από τα όσα προσφέρει στο ιστορική αγορά η πολιτική μας ομάδα. Επομένως, ε, θα στηρίξει τι προσπάθειες του κ. Μπαρνιέ, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικότερα όσον αφορά το ότι θα πρέπει να υπάρχει καταλεπτό, εντελεχώ, παρακολούθηση ε, των επιδόσεων κατομμυρών για τη μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο των ε, οδηγιών και θα πρέπει αυτό να γίνει και για να βοηθήσουμε και την εκτέλεση αυτών των νομοθετημάτων, την εφαρμογή του αλλά και να γίνονται και οι αντίστοιχε καταγγελίε, διαρκή η Το να κατονομάζει κανεί τον ένοχο είναι σκληρό, αλλά πολλέ φορέ χρειάζεται και γι' αυτό το λόγο θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει κάτι σαν ε, ένα νομοθέτημα, σαν πρόγραμμα και έτσι να βοηθήσουμε την ολοκλήρωση τη αγορά. Οπότε να δίνουμε προτεραιότητα σε κάποια μέτρα για να ολοκληρωθεί η ψηφιακή εσωτερική αγορά και επίσης να έχουμε υψηλή ταχύτητα στις συναλλαγές των διασυνοριακών ε, πληρωμών και συναλλαγών και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά τα μέτρα να γίνονται με τρόπο διάφανο και αυτό να γίνει, να γίνει γρήγορα. Πάντως, με την επέτειο που κάνουμε ε, όσον αφορά τον εορτασμό αυτήν την ιστορία αγορά είναι το διαμάντιστο στο στέμα στην ιστορία αγορά v Πράγματι θα εορτάσουμε σύντομα τα 20 γενέθλια της εσωτερικής αγοράς, της ενιαίας αγοράς και θα συμφωνήσω με τις απόψεις του κυρίου Μπουσουτήλ ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα ωφέλη της ενιαίας αγοράς για τους πολίτες μεν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειες για την σωστότερη μεταφορά των οδηγιών και των νομοθετικών ρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο. Έτσι μόνο θα υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις, έτσι θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που του δίδει η ιστοσελίδα, το Solvit και άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και στην δική μου χώρα, στη Σλοβακία, η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τους πολίτες για τις δυνατότητες των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά και που μερικές φορές όμως δεν σέβονται τους κοινοτικούς ε, ε, ορισμούς και νομικές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερα στον τομέα του ε, χείριου κρέατος, ε, υπάρχουν προβλήματα στον τομέα της υγιεινής, όχι μόνο στη δική μου χώρα, στα τρόφιμα ε, και στην Πολωνία υπήρξαν κάποια προϊόντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για ζωοτροφές τα οποία αρχικά έπρεπε να χρησιμοποιηθούν στα δημόσια έργα. Και ξέρουμε επίσης ότι και πουλερικά από τη Γαλλία ε, έγιναν αντικείμενο εξαγωγής σε χώρες όπως η Σλοβακία ε, και τα κρέατα αυτά όμως δεν έπρεπε να μπορούν να κυκλοφορήσουν γιατί ε, δημιουργούσαν προβλήματα υγείας. Το ίδιο επίσης ε, και με κουτιά δημητριακών για πρωινό που περιελάμβαναν ουσίες οι οποίες οδηγούσαν σε τάσεις έμετου. Γενικά όλα αυτά είναι θα έλεγα οι αποδείξεις που πρέπει να μας οδηγήσουμε στη σωστή πιστοποίηση των προϊόντων και την προστασία των πολιτών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα εγώ να, να πω καλά λόγια θα έλεγα για την ενία αγορά αφηρημένα Νομίζω ότι η εσωτερική αγορά και η οικονομική πολιτική μας γενικά πρέπει να έχει σαν στόχο τη λήψη μέτρων προς όφελος των πολιτών. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι δυστυχώς σε αυτή τη φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα, κακές συνθήκες εργασίας και μεγάλη έλλειψη θέσεων απασχόλησης. Συνεπώς ε, δεν ξέρω αν είναι σωστή η αντίληψη ότι η εσωτερική αγορά ε, πράγματι είναι το καλύτερο μέσο για την οικονομική ανάπτυξη. Βέβαια είναι ένα μέσο και αυτό το οποίο απαιτείται μια νέα μορφή οικονομική πολιτικής η οποία να είναι πράσινη και η οποία να βάζει σαν βασικό στόχο του συστήματος τον πολίτη θα πρέπει να διασφαλίζεται η άμεση επαφή των ενδιαφερομένων με αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτούς οι οποίοι διακανονίζουν θα έλεγα και ρυθμίζουν την εσωτερική αγορά αλλά για να το πετύχουμε αυτό πολλά μένει να γίνουν ακόμα γιατί δυστυχώς έχουν υπάρξει και πάρα πολλά αρνητικά μέχρι τώρα. Τα μέτρα πρέπει να στηρίζουν τους πολίτες, πρέπει να στηρίζουν το περιβάλλον και όχι τις επιχειρήσεις όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Δεν θα πρέπει να οικοδομούμε τύχη ανάμεσα στους διαφορετικούς τομείς και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις ανησυχίες των φτωχότερων Ευρωπαίων οι οποίοι σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να πάρουν τη βοήθεια που θέλουν. Πριν από 20 χρόνια ξεκίνησε η εσωτερική αγορά και βεβαίως κάποια πλεονεκτήματα είναι φανερά και σημαντικά για τους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχουν όμως ε, σήμερα μέσω των νέων προτάσεων καινούριες δυνατότητες για να εντοπιστούν και να ξεπεραστούν τα συνεχιζόμενα προβλήματα, αυτά που δεν έχουν ξεπεραστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουμε σε μέσα, σε προσωπικό και δεν είμαι πεπισμένος ότι σήμερα η νέα αυτή η υπηρεσία που ιδρύεται θα βοηθήσει στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά. Είδαμε ότι η οικονομική κρίση μαστίζει τις χώρες της Ευρώπης και δεν έχω την εντύπωση ότι η εσωτερική αγορά μας προστατεύει από όλα τα κακά. Οι συγκεκριμένες θέσεις της Αυστρίας ε, για το θέμα αυτό είναι γνωστό. Είδατε πολύ πρόσφατα στο άρθρο της Frankfurt Allgemeine που αναφέρεται στο θέμα αυτό των πλέον εκτιμάτων από την εσωτερική αγορά ότι κατασκευαστικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και βλέπουμε ότι οι Ευρωπαίοι ε, πολίτες σήμερα βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με έναν σφοδρό ανταγωνισμό όσον αφορά τα ε, εισοδήματά τους και τις πληρωμές τους και ότι βλέπουμε ότι σήμερα αυτή η οικονομική κρίση χρησιμοποιείται για να πλήξει τους εργαζόμενους. και θέλω πρώτα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπάλτα για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, συμμερίζομαι την προτεραιότητα την οποία αναγνωρίζει ο κύριος Μπουσουτήλ και τους στόχους της έκθεσης του και ελπίζω το σώμα να υιοθετήσει την έκθεση αυτή με μεγάλη πλειοψηφία έτσι ώστε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς μια στρατηγική αγοράς για την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης. Αυτό θα επιτρέψει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Πράγματι τα τελευταία αποτελέσματα του πλαισίου αξιολόγησης απέδειξε ότι τα κράτη-μέλη όλο και λιγότερο ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη μεταφορά των ευρωπαϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων. Γι' αυτό τον λόγο συμφωνώ με τον κύριο Μπουσούτιλ για την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δύναμη ισχύς και ευελιξία για την προώθηση και την εκκίνηση των διαδικασιών προσφυγής επί παραβάση και παραβιάση αναγνωρίζοντας βέβαια και τον ρόλο του Solvit Έχω κάποιες επιφυλάξεις για τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που έχουν σχέση τον σεβασμό την αρχή της επικουρικότητας στην περίπτωση κατά την οποία η νομική βάση του Solvit γίνει ιδιαίτερο δίσκαμπτη. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά κάθε είδος λύσης με βασικό στόχο να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα αυτής της ιστοσελίδας χωρίς να δημιουργούνται νομικά προβλήματα. Υπενθυμίζω τελικά ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έχει αναπροσδιορίσει σε βάθος το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδίδοντας του ουσιαστικές εξουσίες και επιτρέποντάς του να αναθεωρήσει την κοινοτική νομοθεσία. Είναι λοιπόν βασικό για να υπάρξει μια σωστή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ε, τα συμπεράσματα του πλαισίου αξιολόγησης να αναλυθούν σωστά στα πλαίσια του διαφθρωτικού διαλόγου ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών. Για τρία λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, την προηγούμενη εβδομάδα πήρα τον λόγο σε έναν ε, οργανισμό γαλλογερμανικής ε, συνεργασίας και μίλησα για τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς λέγοντας ότι σήμερα η εσωτερική αγορά είναι κάτι το αυτονόητο έτσι την καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να μην δημιουργήσουμε νέους φραγμούς, νέα εμπόδια, όπως προσπάθησαν να κάνουν η γερμανική και η γαλλική κυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να διευκολύνουμε την κινητικότητα των ε, πολιτών, των ε, αγαθών και βεβαίως εργαλεία όπως το Solvit και άλλα που σήμερα υπάρχουν είναι πάρα πολύ σημαντικά για να διαπιστώσουμε αν πραγματικά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θέλουν να υιοθετήσουν ευρωπαϊκή νομοθεσία και αν όπως συμφώνησε το Συμβούλιο αυτά θα υλοποιηθούν. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει μία κατηγορία πολιτών που εφολούνται μόνο από αυτήν την κινητικότητα, από αυτά τα μέτρα. Επιθυμούμε να βρεθεί μία συγκρίσιμη αξιολόγηση η οποία να δείχνει πραγματικά τα αποτελέσματα των κρατών μελών. Και σήμερα βλέπουμε παραδείγματος χάρη το Βέλγιο βρίσκεται σε πολύ κακή θέση σε αυτήν την αξιολόγηση. Ο κύριος Πουζουτήλ κάνει κάποιες προτάσεις οι οποίες θα βελτιώσουν αυτήν την δυνατότητα αξιολόγησης. Και την δυνατότητα σύγκρισης των στοιχείων. Εδώ βλέπουμε παραδείγματο χάρη στο άρθρο 18, στο άρθρο 24, στο άρθρο 21, όπως παραδείγματο χάρη ε, την δυνατότητα καλύτερης, ταχύτερης εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, της δυνατότητα ε, μιας πραγματικής σύγκρισης. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εσωτερική αγορά να συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Εγώ άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Χατζημαρκάκη και θεωρώ ότι ήδη οι υπάρχουσες νομοθεσίες οι οποίες έχουν ε, μεταφερθεί και δεν εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται σωστά, όντως είναι το πρώτο που θα πρέπει να μας αντιμετωπίσει και να μας απασχολήσει. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι διαδικασίες οι οποίες προστατεύουν τους εργαζόμενους, την κοινωνική πλευρά αυτών των ε, νομοθετικών κυμάτων θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αν ναι ή όχι εφαρμόζονται. Εμείς είμαστε πραγματικά σε μια καλή θα έλεγα παράδοση σε αυτή την κοινωνική συνεργασία και θα αναφερθώ εδώ στον Ζακ Ντελόρ, πρώην συναδελφό μας, ο οποίος έλεγε ότι η εσωτερική αγορά βασίζεται σε τρεις αρχές, την αλληλεγγύη, την ε, συνεργασία και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον προσέστηκε αυτή η έκθεση, διότι με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε με συγκεκριμένη μέθοδο πόσο βοηθάει την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, η ιστορική αγορά. Πώς θα βρούμε τη διέξοδο από αυτή την κρίση. Είναι πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον. Όμως θα πρέπει να μην τα βλέπουμε όλα μόνο μέσα από το πρίσμα του, του, κεφαλαίου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη οικονομική και κοινωνική των περιφερειακών χωρών της Ευρώπης και των λαών τους, διότι αυτοί που σήμερα στη συγκυρία της κρίσης αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ε, δυσκολίες. Έχουμε μια ε, υπερευαισθησία, είναι, είναι ευάλωτες αυτές οι χώρες σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς ε, ιδιωτικοποιήσεις, απορρίθμιση που γίνεται και πάρα πολλέ χώρε, αυτές που είναι πιο ευάλωτες, έχουν ε, τσακίσει τον παραγωγό του ιστό με τέτοια μέτρα και με κάποιες εισαγωγέ ε, όπως τα ίδια διατροφέ, και στην ε, ενέργεια και έτσι εξαρτώνται πάρα πάρα πολύ από το εξωτερικό. Άρα τι θα γίνει, τι, τι, τι συνέπεια, τι, τι σημασία έχει η εσωτερική αγορά ε, για τη χώρα μας, την Πορτογαλία, για τι ΜΜΕ, για όλες αυτές τις εργασίες που χάθηκαν, για τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη, φτώχεια, το πόσο επεκτείνεται ε, η ευάλωτη θέση απασχόλησης γιατί έχουμε στις ασφάλειες τα ταχυδρομεία, όλες αυτές τις δικοποίησεις σε αυτούς τους ευαίσθητους τομείς. Οπότε ακριβώς ε, από πλευρά σωστικής αγοράς αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μπορεί κάποιος να έχει ελευθερία διακίνησης ε, προσώπων αλλά και εμπορευμάτων θα πρέπει επομένω με τι ελευθερίε κατοχυρωμένε και τα δικαιώματα των εργαζομένων να αντιμετωπίσουν αυτέ τι πολιτικέ οι εργαζόμενοι. την κυρία να Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπουζουτήλ για την ε, έκθεσή του, όχι μόνο διότι πραγματικά είναι πολύ ορθές οι προτάσεις του, αλλά γιατί κυρίως θα μας βοηθήσουν να εργαστούμε πιο αποτελεσματικά, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Περισσότερη διαφάνεια είναι απαραίτητη στην εσωτερική αγορά για να μπορέσουμε και εμείς να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Συμφωνώ απολύτως με τους συναδέλφους που είπαν ότι πρόκειται για μια επιτυχής ε, ιστορία αυτή η οποία διέπει την εσωτερική αγορά. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά η εσωτερική αγορά δεν είναι μια πλήρης επιτυχία. Έχει πολλά πλεονεκτήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό όμως που θέλουμε εμείς είναι όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την αγορά να μπορούν να υποφεληθούν από τις επιτυχίες. Η ιδέα λοιπόν ενός πίνακα αποτελεσμάτων είναι κάτι το πολύ θετικό. Θα πρέπει όμως οπωσδήποτε να είμαστε προσεκτικοί και δεν μπορούμε να ε, παραφηθούμε μόνο στη δημιουργία αυτών των πινάκων αποτελεσμάτων. Πρέπει να δούμε πού χρειάζεται κινητοποίηση των δυνάμεων, πού υπάρχουν αδυναμίες και πού υπάρχουν ε, λανθασμένες ε, κινήσεις. Η έκθεση δείχνει ακριβώς το τι πρέπει ακόμα να κάνουμε, ότι δεν θα πρέπει να χαθούμε στις λεπτομέρειες και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κλείσουμε τα μάτια στα σοβαρά προβλήματα και να ασχολούμαστε μόνο με λεπτομέρειες. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω ιδιαίτερα μία πτυχή ε, αυτό που ήθελα να πω για να σας δείξω ότι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα στην εσωτερική αγορά. Η ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί για τα μεγάλα έργα που αποτελούν περίπου το 20% του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εσωτερικού προϊόντος. Διαπιστώνουμε σήμερα ότι περιέχουν πολύ δύσκολες διακητικές ε, διαδικασίες. Θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, θα πρέπει να γίνουν πιο απλές και πιο ελαφρές οι διαδικασίες. Θεωρώ ότι όντως έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να δούμε η εφαρμογή αυτή της Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, με ποιον, τρόπο γίνεται από τα κράτη-μέλη έλλειψη διαφάνειας, αλλά και κάποιες συγκεκριμένες δράσεις επιτόπου, έτσι ώστε η μεταφορά αυτής της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας να είναι πιο αποτελεσματική. Θα πρέπει να αποφύγουμε επικαλύψεις, θα πρέπει με μεγαλύτερη ταχύτητα να μεταφέρετε το δίκαιο που ακόμα δεν έχει μεταφερθεί, γιατί από αυτό εξαρτάται και η ασφάλεια και η ανάπτυξη, αλλά και οι θέσεις εργασίας. Οι πίνακες αποτελεσμάτων δεν πρόκειται να επιλύσουν όλα τα προβλήματα. Δεν αρκούν σε καμία περίπτωση, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πολλά από τα κράτη-μέλη πολύ περισσότερο. γιατί ακόμα όλα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Επίτροπε, είμαστε όλοι πεπισμένοι για τη σημασία που έχει η εσωτερική αγορά για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Έπαιξε τα τελευταία 20 χρόνια η ενιαία αγορά ένα χαρακτηριστικό της ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί η δυνατότητα ανάπτυξης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως μέσω της έννοιας αγοράς. Συμφωνούμε με το ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε κάποια από τα θέματα που ήδη έχουν τεθεί βέβαια από τους προλαλήσαντες. Ο πραγματικός εχθρός της ενίας αγοράς είναι φυσικά η κρίση. Αυτή αμφισβητεί την εικόνα που έχει αποκτήσει η ενιαία αγορά στα μάτια των πολιτών. Είναι κάτι το οποίο μειώνει την προστιθέμενη αξία της αγοράς αυτής. Πρέπει λοιπόν να εμείνουμε στην ανάπτυξη, στην ιδέα της ανάπτυξης, γιατί χωρίς την ανάπτυξη η προσπάθειά μας για την εσωτερική αγορά καθίσταται πολύ δυσκολότερη. Η διαδικασία κρίσης την οποία βιώνουν οι χώρες μας παράγει και άλλη μία αρνητική πλευρά δίδει δικαιολογίες αν θέλετε, αστήρικτες πάντα σε ορισμένες χώρες έτσι ώστε να εφαρμόζουν με στρεβλό τρόπο ή διαφοροποιούμενο τρόπο αυτά που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δημιουργούνται δύο προβλήματα. Πρώτον, καθυστέρησης της πληρωμές από πλευράς των κρατών μελών που δεν είναι θέμα γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά είναι λάθος πολιτικών στόχων. Και δεύτερον, η σωστή αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των πληρωμών. Πολλές φορές ε, δημιουργούνται προσπάθειες στην κατανόηση της μορφής της παρέμβασης στα πλαίσια της αξιολόγησης ε, ε, βγαίνουν ορισμένα συμπεράσματα με βάση τον μέσο όρο, αλλά ε, με τα επιμέρους στοιχεία βλέπει κανείς ότι έχει μια Ευρώπη η οποία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα τα οποία έχει, τις πιστώσεις που έχει στη διάθεσή της, με όχι πολύ διαφανή τρόπο. Λοιπόν, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να ενισχυθούν. Το ίδιο και οι κυρώσει σχετικά με την μη σωστή εφαρμογή ή με την μεγάλη καθυστέρηση εφαρμογή των συμπεφωνημένων. Να πω εδώ ότι και το Solvit είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ευαίσθητο θέμα βέβαια το να αναζητήσουμε τη νομική βάση σωστά, αλλά έχει αποδείξει θετικά πράγματα το Solvit, δεν πρέπει να το εκαταλείψουμε. Να πω κάτι στον εισηγητή ότι σε αυτή τη φάση αντιμετωπίζουμε επιπλέον δυσκολίες και δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο έχει γίνει η πρόταση ενός τρίτου του εισαγγελέως εισαγωγικά για την εσωτερική αγορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει περαιτέρω δυσκολίες, περαιτέρω καθυστερήσεις και μια τέτοια πρόταση φοβάμαι δεν έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σήμερα διαπιστώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μας πλήττει η οικονομική κρίση. Η εσωτερική αγορά είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, καθότι αποτελεί το εργαλείο το πιο σημαντικό που έχουμε στα χέρια μας. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε και την Επιτροπή αλλά και τις Εθνικές Αρχές, οι οποίες θα πρέπει να δεσμευτούν περισσότερο έτσι ώστε οι οδηγίες, τα νομοθετικά κείμενα εγκαίρως και εντός των προθεσμιών να μεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη διαφάνεια. Θα πρέπει να ενημερώνεται και ο πολίτης και οι επιχειρήσεις. Και σε αυτό θα, το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω εξαιρετικά τον κύριο Μπουζουτήλ για την εξαιρετική του έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ο λόγος και πάλι στον κύριο Ανδρέα Σουάπ για τρία λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι εκπλήσωμαι όταν ακούω κάποιους συναδέλφους. Ο κύριος Κούσταυσον από τους αριστερούς δεν είναι εδώ, λέγοντας ότι η εσωτερική αγορά έριξε πολύ κόσμο στην φτώχεια, αυτό πραγματικά με εκπλήσει, με ανησυχεί. Στη δική μου παραδείγματο χάρη εκλογική επικράτεια όπου δεν υπάρχουν ε, εκλογική περιφέρεια όπου δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, βλέπω πραγματικά ότι οι πολίτες εποφελούνται από την εσωτερική αγορά. Και αν κοιτάξω τη δική μου περιφέρεια, διαπιστώνω ότι αυτά τα λεγόμενα δεν είναι ορθά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της μεταφοράς ε, της οδηγίας στην Γερμανία, όπως είπε η κυρία Βάιλ, κάτι που γίνεται πολλές φορές καθυστερημένα. Εμείς θέλουμε η οδηγία η οποία έχει υιοθετηθεί εδώ με δημοκρατικό τρόπο και με την συμφωνία του Συμβουλίου να εφαρμοστεί παντού και στη Γερμανία. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα πραγματικά να ακουστεί με μεγάλη σαφήνεια. Στην έκθεση Μπουζουτήλ αναφέρεται η ανάγκη για περισσότερα νομοθετικά κείμενα, περισσότερους κανονισμούς και οδηγίες. Διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία. Όσον αφορά τον κανονισμό υπάρχει βεβαίως μια δυνατότητα όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των νομοθετικών κειμένων και θα πρέπει σίγουρα στο μέλλον να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί γιατί βλέπουμε ότι το έλλειμμα μεταφοράς είναι κάτι που θα πρέπει να το μειώσουμε με δραστικό τρόπο. Και ξέρω ότι ο κύριος Μπαρνιέ, όπως και η πολιτική ομάδα του ΕΛΚ, σαφώς και επιθυμούν να γίνει μία συζήτηση όσον αφορά την θέση των οδηγιών και τη θέση των κανονισμών. Κυρία για λεπτά παρακαλώ. Øh, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πριν από πολλά χρόνια που ήμουν μικρή, καθόλου δεν με ενθουσίαζε η ιδέα της ενιαίας αγοράς, γιατί εγώ θεωρούσα ότι θα φερθούν μόνο οι καπιταλιστές και όχι οι λαοί. Συνήλθα όμως ευτυχώς και άλλαξα γνώμη. Είδα τι θα πει εσωτερική αγορά στην πράξη. Και σήμερα πρόκειται για μια ατμομηχανία συνεργασίας. Πρόκειται για συμβολή στην ανάπτυξη, στην ευημερία, στην απασχόληση. Πάντως, επίσης είναι σημαντικό να συνεχίσει να παίζει η ιστορική αγορά αυτό το ρόλο και στο μέλλον γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ιστορική αγορά να συνεχίσει να λειτουργεί καλύτερα από όσο λειτουργήσε στο παρελθόν. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει το εκπρόσωπο του Συμβουλίου να ακούσει τη σύντησή μα, διότι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό είναι τα κράτη-μέλη να αντιληφθούν ότι έχουν ευθύνη τεραστία να εξασφαλίσουν ότι η θεσπιζομένη νομοθεσία εφαρμόζεται ορθά. Πάρε πολύ καλά τα είπε ο κύριος Μπουσούτιλ. Δεν τα πάνε πολύ καλά οι χώρες μας. Αλλά αν τα πήγαιναν όπως τα πάει η Μάλτα, τότε όντως θα ήταν μια χαρά η εσωτερική αγορά, οπότε τελικά είναι θέμα πολιτική βούλη των κρατών μελών. Αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί. Θα πρέπει να τα καταφέρουμε εμεί καλύτερα. Γιατί εάν δεν τα καταφέρουμε καλύτερα, τότε θα χάσουμε την υποστήριξη των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων. Ακόμα και σήμερα κοροϊδεύουμε τους αγρότες με τα καινούρια κλουβιά για τα κοτόπουλα τις οτόκες όρνητες γιατί μπορούμε να έχουμε αυγά από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής όμως ο κόσμος μπορεί να στηριχθεί στην αξιοπιστία, στην ασφάλεια της εσωτερικής αγοράς. Να πώς λειτουργεί η εσωτερική αγορά και εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε οι εργαζόμενοι, οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους, γιατί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν θεμητούς όρους ανταγωνισμού οι αρχές, τότε ε, ότι αυτοί μπορούν να λάβουν κάποια κάλυψη. Γι' αυτό και εμείς θεωρούμε ότι αυτός ο πίνακας επιδόσεων και αποτελεσμάτων είναι πάρα πολύ σωστή ιδέα. Επίση, συμφωνώ και με την ιδέα του κ. Μπουσούτιλ σε σχέση με αυτή τη διαδικασία fast track, τη συνοπτική διαδικασία όσον αφορά εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία θα πρέπει κάτι να κάνουν γιατί δεν προχωρούν όσο πρέπει σήμερα και βλέπουμε το πώς μπορεί να έχουμε μια task force η οποία να πηγαίνει γύρω-γύρω στις πρωτεύουσες να βοηθάει στην εφαρμογή της Μεταφορά του κοινοτικού υγείου στην εσωτερική ενωμή τάξη. Ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Έχετε δίκιο κύριε Μπουσούτελ. Και την επόμενη 20 ετία μπορούμε να ισχυριζόμεθα ότι η ιστορική είναι για τους πολίτες και όχι αντίστροφα. Την αίθουσα, οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω τον ε, κύριο Ρέπο να πάρει το λόγο. Για τρία λεπτά παρακαλώ. Ε, ε, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κοινωνική ειρήνη και η κοινωνική δικαιοσύνη που έχουμε πετύχει ήταν τα θεμέλια για την ευρωπαϊκή συνεργασία. Όμως, κατέθεσαν εφικτά με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, γιατί η Ευρώπη δίνει πλειάδα ευκαιριών. Όμως, ελοχεύει ένας κίνδυνος να χάσουμε, να υπονομεύσουμε αυτές τις ευκαιρίες. Γι' αυτό το λόγο και είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση γιατί τοποθετείται στο πρόβλημα της ε, μεταφοράς του ιστορικό δίκαιο των ευρωπαϊκών οδηγιών. Γιατί είναι πάρα πολλές οι οδηγίες που δεν το κάνουν αυτό όπως θα έπρεπε. Κανονισμούς και οδηγίες δεν τηρούν τις προθεσμίες που τάσσονται για αυτή την ε, ενσωμάτωση στο ιστορικό δίκαιο. Και κυρίως ε, τα προβλήματα υπάρχουν στην περιβαλλοντική νομοθεσία και την φορολογική νομοθεσία. Αυτή επομένως η προβληματική κατάσταση παραβλάβεται σήμερα των κρατών μελών που βραδύνουν να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, αλλά παραβλέπεται και τα συμφέροντα των υπολείπων κρατών μελών. Γιατί αν θέλουμε αλληλεγγύη που θα βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη, τότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η μεταφορά θα γίνεται ε, ταχύτερα. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να βρουν την πολιτική βούληση για την ε, εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μόνο έτσι η Ένωση να θα πετύχει τους στόχους της στρατηγικής για το 2020. Ας πούμε για τα θέματα τα ενεργειακά, τους ενεργειακούς πόρους, υποτελεσματική χρήση της ενέργειας, γιατί επίσης ε, το πρόβλημα αυτό το οποίο τώρα συζητούμε υπονομεύει την αξιοπιστή Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανταγωνιστικότητά της και ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων. Πώς να ζητάμε από τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν στην επίτευξη των κοινών στόχων εάν εκείνοι επιλαμβάνουν τις αποφάσεις εάν τα ίδια τα κράτη-μέλη δεν είναι πρόθυμα να πράξουν το ίδιο το οποίο απαιτούν. Η κοινωνική νομοθεσία αποσκοπεί στο να δημιουργήσει καλύτερο κλίμα για τις ΜΜΕ αλλά και καλύτερου όρου για του καταναλωτέ. Όμω αυτό δεν θα γίνει αν δεν υπάρχει κοινή νομοθεσία και αν δεν υπάρχει κατάλληλη προσαρμογή, επικαιροποίηση αυτή τη νομοθεσία και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε, να παρέμβουμε όταν κάποια κρατημέλη με τι ενέργειε του δεν τηρούν τι δεσμεύσει του για αυτού, του κοινού κανόνε και αν δεν κάνουμε κάτι όσον αφορά αυτέ τι παραβάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, τη παραβιάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, τότε οδηγούμεθα στην κατάτμιση τη εσωτερική αγορά γιατί περί αυτού πρόκειται. Να, πώς οδηγήκαμε στην σημερινή κρίση. Είναι και θέμα ηθικό. Θα πρέπει όλα τα κρατημέλη να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να μπορέσουμε να τις αποτύχουμε. τους κοινούς μας στόχους. παρακαλώ, για δυόμιση λεπτά. Ε, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μπουσούτιλ για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του. Η ενιαία αγορά είναι ένα πεδίο στα πλαίσια του οποίου όλα τα κράτη-μέλη χωρίς καμία εξαίρεση συμφωνούν ότι αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια ουσιαστική θα έλεγα δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Για τη σωστή λειτουργία όμως της ενιαίας αγοράς πρέπει τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν στην ομοθεσία τους τις ευρωπαϊκές νομικές ρυθμίσεις. Έχει υπάρξει μια κάποια πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες θα έλεγα έχουν μείνει αρκετά πίσω. Θα πρέπει στα πλαίσια της μεταφοράς αυτής του ευρωπαϊκού δικαίου στις χώρες μέλη να υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το πρώτο εμπόδιο το οποίο διαπιστώνεται είναι ε, στη στιγμή της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Όταν γίνονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αντίθεση, για να μην πω αντίσταση ορισμένων κρατών μελών, στην ίδια της, την ιδέα της δημιουργίας των λεγόμενων ε, πινάκων αποτελεσμάτων, η συγκρισιμότητα, αξιολόγησης, που επιτρέπουν να διαπιστώνουμε σε ποιο βαθμό έχουμε περάσει στην απαιτούμενη εναρμόνιση. Παρ' όλα αυτά οι πίνακες αυτοί είναι το πρώτο βήμα έτσι ώστε να υπάρξει τακτική παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο βελτιώνονται τα θέματα στον τομέα της μεταφοράς της νομοθετικής. Πρέπει λοιπόν η αδίποτε ε, νομική ευρωπαϊκή πράξη να εφαρμόζεται σωστά. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Όπως ευχαριστώ και το φίλο μου, το Σιμών Μπουσουτήλ, για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. Είχα ετοιμάσει μία άλλη ομιλία, αγαπητέ Σιμών. Αλλά δυστυχώς θα πω άλλα πράγματα και θα πω άλλα πράγματα διότι ήρθε σε γνώση μου αυτή εδώ η τροπολογία και αυτή εδώ η τροπολογία αλλάζει τελείως το κλίμα αλλάζει τελείως την έκθεση. στην ελλάδα έχουμε ένα τραγούδι πάρα πολύ γνωστό το οποίο λέει πως ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο. το θυμάμαι αυτό το τραγούδι τώρα διότι η δική σου έκθεση αγαπητέ σιμών ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. ήταν ένα κείμενο ευρείας κοινή αποδοχής. στην επιτροπή ψηφίστηκε ομόφωνα. δεν θα τελειώσουμε όμως καλά. και δεν θα τελειώσουμε όμως καλά διότι η υπόθεση της εσωτερικής αγοράς και ειδικά του πίνακα των αποτελεσμάτων του λεγόμενου scoreboard δεν αφορά αριθμούς αφορά ανθρώπους αφορά τους ευρωπαίους πολίτες και μάλιστα αφορά τους ευρωπαίους πολίτες σε καιρό κρίσης. όταν το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο συζητά προβληματίζεται νομοθετεί το κάνει για τους ευρωπαίους πολίτες και το κάνει όχι in vitro αλλά προβληματίζεται και νομοθετεί in vivo. η ίδια η ζωή είναι που μας ενδιαφέρει έτσι λοιπόν ο πίνακας των αποτελεσμάτων ξέρουμε ότι αποτυπώνει εάν κάθε χώρα μέλος μεταφέρει την ευρωπαϊκή νομοθεσία σωστά και την εφαρμόζει σωστά στην περιοχή του. ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν κράτη μέλη που καθυστερούν. συμφωνούμε όλοι ότι αυτά τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεχθούν επιπλήξεις θα πρέπει ενδεχομένως να δεχθούν και ποινές. πριν όμως φτάσουμε στην ποινή θα πρέπει να εξετάσουμε γιατί αυτά τα κράτη καθυστερούν. τι φταίει ακριβώς; το γεγονός ότι οι μισές εκρεμείς υποθέσεις αφορούν τη φορολογία και το περιβάλλον λέει πάρα πολλά πράγματα γιατί βρισκόμαστε στον καιρό που συζητάμε για την οικονομική και την νομισματική ένωση και βλέπουμε πως όταν αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν έχουμε προβλήματα και έχουμε κρίση στην ευρώπη και έχουμε ένα ευρώ να απειλείται. και έρχεται λοιπόν αυτή εδώ η τροπολογία η οποία λέει ούτε λίγο ούτε πολύ να φτιάξουμε έναν εισαγγελέα να κατασκευάσουμε έναν εισαγγελέα άλλο ένα σώμα ελεγκτικό και σώμα που θα αποδίδει ποινές για να βάλουν μυαλό τα κράτη μέλη. φοβούμαι αγαπητέ σιμών φίλε σιμών και αγαπητέ επίτροπε ότι με τέτοιου τύπου ενέργειες δεν πάει μπροστά η ευρώπη και δεν γίνεται ελκυστική η εσωτερική αγορά. παρακαλώ πάρα πολύ να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τελειώνω κυρία πρόεδρε το θέμα των κινήτρων και των ποινών γιατί αντικατοπτρίζουν και αντιλήψεις. εμείς ως σοσιαλιστές και δημοκράτες είμαστε υπέρ των κινήτρων. δεν πιστεύουμε ότι το epp είναι μόνον υπέρ των ποινών. ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ράπτη. Η κυρία Μπάστος δεν είναι στην αίθουσα, όπως επίσης και η κυρία Χέρτσοκ, Οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω τον ε, κύριο Χάρμπορ να πάρει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, με μεγάλη μου χαρά συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Βέβαια ήρθα λίγο πιο αργά από όσο περίμενα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με αφήσατε να λάβω το λόγο και επίση με συμπαθά και ο κύριο Σάιμον Μπουσούτελ. Πάντω τον συγχαρητήρια για την εισήγησή του και ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο για τη δική του απάντηση. Όμω, μια που είμαι πρόεδρο τη αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, θέλω να σα πω ότι χαίρομαι που είναι τόσοι συνάδελφοι εδώ να στηρίξουν αυτή την έκθεση και φυσικά, όπως είπε και η κυρία Ράπτη, δεν μπορούμε όλοι να συμφωνούμε σε όλα. Όμω νομίζω ότι η εντελεχής ανάλυση των θεμάτων ε, που διεξέρχεται αυτή η έκθεση δείχνει το πόσο ασχολούμε, θα διεξέρουμε τα θέματα στην ε, ε, Επιτροπή μα. Και ξέρω επίσης ότι, κύριε Επίτροπε, θα πάρετε το, το, το θέμα στα σοβαρά, όπως είπατε στην αρχή. Τους άκουσα, ε, όσους άκουσα, δεν τους άκουσα όλους, γι' αυτό δεν ξέρω εάν θα ξαναπώ τα ίδια πράγματα. Πάντως, θέλω να σας πω τα εξής ούτως ώστε να επισημάνω δύο συγκεκριμένα θεματάκια. Το είπε και η κυρία σχετικά με τις ε, παραβάσεις του κοινωτικού δικαίου, όμως ε, θέλω να τονίσω κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου αποτελεί την εξέλιξη της εποπτείας μας και της εξολόγησής μας για το τι πετυχαίνει και πώς λειτουργεί η ιστορική αγορά, διότι ακόμα έχουμε πολλές χαμένες ευκαιρίες. Και ο κύριο Μπόκλεστάιν σε μια ετήσια έκθεση είχε πει ότι η ιστορική αγορά είναι σαν μια Φεράρι η οποία όμως την οδηγεί κάποιος με την δευτέρα ταχύτητα. Επομένως, δεν μπορεί βέβαια να φτάσει πολύ ψηλή ταχύτητα. Πάντω ε, είναι γερό αυτοκίνητο. Από την άλλη μεριά, την, αυτή, αυτή η Ferrari που έχουμε εμεί εδώ είναι Ferrari που μπορεί να την οδηγήσει ο καθένα. Και το πρόβλημα το οποίο τελικά έχουμε είναι ότι δεν ξέρουμε πόσε ακόμα επιπλέον χαμένε ευκαιρίε υπάρχουν γιατί έχουν προσπαθήσει κάποιε επιχειρήσει να προωθήσουν αγαθά, εμπορεύματα, υπηρεσίε κάπου και με θεμητό τρόπο και παρόλα αυτά δεν μπορούν να το κάνουν διότι ε, προσκρούν σε πάρα πολλούς φραγμούς. Φραγμούς που αντιμετωπίστηκαν από τα σχετικά νομοθετήματα της νοηδηγίας της υπηρεσίας και αυτά και τελικά τελικά σηκώθηκαν αυτέ οι επιχειρήσει και πήγαν αλλού. Τα μάθησαν και πήγαν αλλού. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε υπολογίσουμε πόσε είναι αυτέ οι χαμένε ευκαιρίε και να δούμε τι γίνεται και με τη στάση των ε, επιχειρήσεων. Το Solvit ε, αυτό το, σημείο, το ενιαίο σημείο επαφής όλα αυτά μας δείχνουν το πόσες χαμένες δυνατότητες υπάρχουν αναξιοποιητές γιατί θα πρέπει να κοιτάξουμε ε, στην έκθεση μια πάρα πολύ μικρή παραγραφή και λέω ότι θα πρέπει να δούμε το ευρωβαρόμετρο τι λέει, τι λέει στην, στην, ετήσιο έλεγχο της ε, διακυβέρνησης. Ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την ετήσια έκθεση του ευρωβαρόμετρου δεν αναφέρεται σχέση με την ιστορική αγορά ότι θα πρέπει να έχουν και κάποια μέτρα συνειδητοποίησης, κάποια μέτρα ε, πληροφόρηση, ούτω ώστε όλοι να ξέρουν τα δικαιώματά τους, να ξέρουν για το σημείο ενιαίο σημείο επαφή. Αλλιώς δεν θα έχουμε ιδέα για το τι κάνουν τα κράτη-μέλη, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ευρωπλατφόρμα, πολύ σωστά πάνε συνάδελφοι, και έτσι να έχουμε μία επωνυμία εμπορική που να τους καλύπτει όλους. Και τελικά η κεντρική ιδέα της έκθεσης είναι να υπάρχουν αυτές οι συνοπτικές διαδικασίες. Ακόμα είμαστε σε πρώιμη φάση για να δούμε πού θα πάει αυτή η ιδέα αλλά υπόσχεται πολλά ιδέα αυτή του κυρίου Μπουσούτη και Εάν κάποιος δεν μπορεί να προωθήσει ένα εμπόρευμα ή μια υπηρεσία γιατί μια κυβέρνηση δεν εφαρμόζει την κοινωνική νομοθεσία, θα πρέπει εντάχει να αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Διότι αν δεν απονέμεται ταχύω δικαιοσύνη, δεν απονέμεται καθόλου δικαιοσύνη. Στην ε, διαδικασία Catch the Eye και θέλω πρώτα να δώσω το λόγο στην κυρία Μαζέη Κουκοβίτς. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Τι. Ε, πρόκειται για την 20η επέτειο τη εσωτερική αγορά. και βρισκόμαστε ει ε, συγκυρία πολύ σκληρή κρίση. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη και τα λαμβάνει η έκθεση του κύριου Μπουστούτ και γι' αυτό και χαιρετίζουμε την ε, παρουσιασή της και θα πρέπει επομένως να δούμε το πώς θα ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας λιγότερο να στρέφουμε επομένω τις δυνατότητές μας για να ανταγωνιστούμε άλλους, άλλους στην διεθνή σκηνή όπως τις χώρες BRICS. Γι' αυτό και θεωρώ ότι κάθε τέτοια νομοθεσία που σε αυτήν την κατεύθυνση είναι θετική για μένα και νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε καλύτερα το, το, το, το, πόσο θα πρέπει να επικοινωνούμε καλύτερα. Και αυτό διότι η οι σχετικέ ιντερνετικέ, οι σχετικέ διαδικτυακέ πύλε υπάρχουν παντού. Όμω τι γίνεται, δεν λειτουργούν καλά αυτέ οι διαδικτυακέ πύλε. Θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με λόγια, με, με, με τον προφορικό λόγο. Και άρα οι ΜΜΕ να γνωρίζουν καλύτερα το τι γίνεται με αυτές τις διακτικές πύλες. Κυρία Μπασέσκου, παρακαλώ. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Piața unică joacă un rol crucial în ieșirea Europei din stat. Η εσωτερική αγορά παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στις ευρωπαϊκές προσπάθειες να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμόζονται πλήρως και εγκαίρως όλες οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια είναι ουσιαστική καθότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ενιαίας αγοράς θα γίνει ισχυρότερο και οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης θα υποφεληθούν από μια τέτοια βελτιωμένη εσωτερική αγορά. Ο πίνακα των αποτελεσμάτων έχει σαν σκοπό να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα κράτη-μέλη. Δυστυχώς οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν επιτευχθεί από τη χώρα μου. Η Ρουμανία θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπαθίες της έτσι ώστε να βελτιώσει τις μεταφορές. Όταν ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούσαμε τις λέξεις ελεύθερο εμπόριο ε, και όχι εσωτερική αγορά. Ήταν κάτι το οποίο βέβαια είχε δημιουργήσει ψευδεστήσεις σε σχέση με την πραγματικότητα. Η, ε, θα έλεγα η σημερινή κατάσταση δυστυχώς οδηγεί στην ελεύθερη μετακίνηση μεν των εργαζομένων, διακίνηση των εργαζομένων, αλλά και στην απώλεια όμως ε, των θέσεων απασχόλησης των ιδίων εργαζομένων. Η πρόταση αυτή στην ουσία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινά άμεσα διαδικασίες επί παραβάση εναντίον χωρών μελών που δεν έχουν μεταφέρει ε, τις ευρωπαϊκές νομιθετικές ρυθμίσεις ε, στην εθνική νομοθετική τάξη. Από το 1973 όταν εμείς ε, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία είχαμε ε, προειδοποιήσει για αυτήν την οργουελική πραγματικότητα την οποία επεφύλασαν στους εργαζομένους οι ευρωκράτες. Η κυρία Τούνουντ Χόχενστάιν. pani przewodnicząca! <clears throat> ten e, scoreboard single market scoreboard Ο πίνακα αποτελεσμάτων τη ενιαία αγορά είναι εξαιρετικά σημαντικό και όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βάλουμε στο κέντρο τη ε, συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στην Ευρώπη και στι χώρε μα. αυτό το πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς. Τα στοιχεία που ε, περιέχει αυτός ο πίνακας θα πρέπει να μας βοηθήσουν. Χρειαζόμαστε και στοιχεία και συγκρίσεις και ανταλλαγή καλών πρακτικών και μελέτες και ερωτηματολόγιο και διαδικτυακές πύλες και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το φόρουμ που είχα προτείνει στην έκθεσή μου πριν από δύο χρόνια το Φόρουμ για την Εσωτερική Αγορά λειτουργήσε με, με εξαιρετικό τρόπο, γι' αυτό και θα ήθελα να διοργανώνουμε κάθε χρόνο κάποιες μέρες ή μία εβδομάδα της εσωτερικής αγοράς. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο η εσωτερική αγορά θα γίνει κατανοητή σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και ζητώ από τον Επίτροπο, τον κύριο Μπαρνιέ, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας, για τις προτάσεις σας. Ε, να ευχαριστήσω κυρίως τον κύριο Σφάμπ γιατί υπογράμισε στην αρχή της παρουσίασής του το ότι όταν να μιλάμε για την ενιαία αγορά μιλάμε για αυτό το απόθεμα ανάπτυξης να πω επίσης και ειδικά στον κύριο Κοφεράτη που αναφέρθηκε στην κρίση σαν βασική απειλή ότι στην αρχή της παρουσίασής μου είπα κάτι το οποίο συναντά και καλύπτει αυτά τα οποία εσείς είπατε. Και το επαναλαμβάνω, στα πλαίσια αυτής της κρίσης, μέσω της εθνικής αναδίπλωσης και της ανόδου του προστατευτισμού, το πρώτο θύμα θα είναι η εσωτερική αγορά. Αν καταστήσουμε αποσπασματική και διακεκομένη την λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω προστατευτικών εθνικιστικών τάσεων δεν θα επιβιώσει η ενιαία αγορά. Για να βγούμε όμως από την κρίση αυτή, αυτή η μεγάλη εσωτερική αγορά απαιτεί περισσότερη ελευθερία, λιγότερο αποσπασματική αντίληψη για να ξαναβρούμε την ανάπτυξη. Έτσι θα συναντήσουμε εκ νέου την ανάπτυξη για να λειτουργήσει σωστά η ενιαία αγορά θα πρέπει να γίνει σωστά κατανοητή. Ο Αλγκόρ είχε πει ότι είναι βασικό να κατανοήσουμε το πού βρίσκονται οι αδυναμίες μας. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τα λάθη μας, τις ανεπάρκειές μας στον τομέα της επικοινωνίας, ε, έτσι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά και γι' αυτό ακριβώς δημιουργούμε αυτούς τους πίνακες αξιολόγησης και να πω επίσης προς τον κύριο Σφάμπ ότι πέραν αυτής της σφαιρικής αν θέλετε πρότασης θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο επιμέρους και να εξετάσουμε κατά περίπτωση το πώς λειτουργεί η νομοθετική ε, αυτή τη στιγμή πλαισίωση της ενίας αγοράς. Ξέρουμε ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες, σαν παράδειγμα, αποκαλύπτει το 40% της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί πάρα πολύ προσεκτικά στα πλαίσια του συνολικού πίνακος να αναλύσουμε επιμέρους όλα τα συστατικά στοιχεία. Όπως έλεγαν και άλλοι συνάδελφοί σας, στην ουσία ο πίνακας αυτός θα είναι σαν ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, θα δείχνει αν θέλετε ποιοι πάνε καλά και ποιοι λιγότερο καλά και κυρίως θα μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε τα κράτη να επιλέξουμε τις σωστές πρακτικές και θα έλεγα προς τον κύριο Σφαμπ πάλι και τον κύριο Στόλογιαν ότι συμφωνώ μαζί τους ότι θα πρέπει να υπάρχουν και οι πίνακες αντιστοιχίες για όλα τα νομικά κείμενα, για όλες ε, τις οδηγίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις σωστές συγκρίσεις. Τώρα για τις ε, διαδικασίες επί παραβάση είμαι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσω τις διαδικασίες αυτές όπως το έχουμε ήδη κάνει για να υποχρεώσουμε τα κράτη να κάνουν αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν. Αλλά πριν φυσικά θα προσπαθήσω να εξαντλήσω κάποιες δυνατότητες χορήγησης κινήτρων, πυθούς και προσπαθώντας να είμαι αντικειμενικός κάποια πράγματα έχουν βελτιωθεί. Χάρη στις πρωτοβουλίες γύρω από το U-Pilot μειώσαμε κατά πολύ τον αριθμό των διαδικασιών επί Θα ήθελα να μειώσουμε επίσης και τις χρονικές διαδικασίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα μακρόχρονες, μεγάλες. Λοιπόν, ανάμεσα στα μέσα που έχουμε για να φέρουμε κοντά τις βεξέλες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις είναι το Solvit. Αυτό το Solvit το πιστεύω πραγματικά. Νομίζω ότι θα τα Solvit σε κάθε κράτος μέλος, όπως είπε και ο κύριος Τοσκάμπος και ο κύριος Όμπεμάγερ, το Solvit θα πρέπει να έχει τα νομικά μέσα τα τεχνικά μέσα και το προσωπικό που απαιτείται σε κάθε χώρα για να λειτουργήσει σωστά. Πολλοί από εσά, όπως και ο κύριος Μπουσούτιλ και η κυρία Ράπτη και η κυρία Τάιλερ αναφέρθηκαν σε αυτήν τη νέα ιδέα του κυρίου Μπουσούτιλ του εισαγγελέως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με αυτή την πρόταση. Θα με καταλάβει εδώ ο κύριος Μπουσούτιλ. Εμείς εργαζόμεθα στα πλαίσια των συνθήκων, είμαστε θεματοφύλακες των συνθήκων και θα πρέπει να αποφύγουμε τις πολλαπλές επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και λειτουργιών. Βέβαια έχετε κάθε δικαίωμα σαν νομοθέτης να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει σωστά τη δουλειά της χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει σαν ρόλο να ελέγχει πολιτικά το τι κάνουμε. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, σας ανήκουμε, συνεργαζόμαστε και με το Συμβούλιο και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Κύριε Μπουσούτιλ, θα πρέπει να ισχυθεί εδώ ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε όλα αυτά τα νομικά κείμενα να εφαρμόζονται σωστά στις χώρες μέλη. Έχουμε κάποιες βασικές ιδέες εδώ τις οποίες θα εξετάσουμε έτσι ώστε σαν παράδειγμα να καθορίσουμε τις κατά προτεραιότητα τομείς και δραστηριότητες. Έχοντας κάνει την προεπιλογή αυτή και έχοντας επιλέξει τους τομείς τους πιο αποτελεσματικούς για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, να έχουμε μια ενισχυμένη εταιρική σχέση με τα κράτη-μέλη και να καταλήξουμε σε επίπεδο ανοχής μηδέν. Αυτό το οποίο στοχεύει και ο κύριος Μπουσούτιλ με την τροπολογία του. Αποφασίσαμε επίσης να προτείνουμε η προσπάθεια αυτή για τη σωστή εφαρμογή της εσωτερικής αγοράς να συμπεριληφθεί σε μια δεσμευτική διαδικασία, νομικά εννοώ το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να μην περιοριστούμε σε μια αξιολόγηση σε επίπεδο αυστηρά δημοσιονομικό, αλλά και σε επίπεδο ανάπτυξης, κάτι το οποίο έχω συζητήσει και με τον συνάδελφο Ρένα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δουλέψουμε σωστά, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στον διάλογο με τις επιχειρήσεις μικρές και μεσές. Να πω και προς τις άλλες συναδέλφους σας ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή η εβδομάδα της εσωτερικής αγοράς, μια ιδέα που γεννήθηκε μετά από την επιτυχία του, του φόρουμ της Κρακοβίας την οποία είχε φανταστεί και η συνάδελφός σας ο Ζακούν. Ε, μέσω και των δικτύων ε, του, μέσω του διαδικτύου, μέσω των κοινωνικών δικτύων επικοινωνίας, όπως και ο κύριος Χάρμπορ το ζήτησε και ο κύριος Σφάμπ και ο συνάδελφός μου ο κύριος Ταγιάννη, θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το διάλογο με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν άμεσα και σωστά το διαδίκτυο και να είναι απόλυτα ενήμεροι σε σχέση με το τι έχουμε κάνει και τι κάνουμε για τη διευκόλυνση του τρόπου εργασίας τους. Να συμφιλιώσουμε τους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εσωτερική αγορά. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε και αυτό είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Μπαλτασάρε λέγοντας ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τα κοινοβούλια των χωρών μελών. Όταν μιλάμε για ελευθερία διακίνησης και εμπορευμάτων και απαντώ εδώ στον κύριο Πάσχα, μιλάμε ακριβώς για την ασφάλεια αυτών των προϊόντων. Κύριε Πάσχα, όταν τα προϊόντα αυτά έρχονται στην εσωτερική αγορά πρέπει να σέβονται ε, τα, τους, τις νομικές ρυθμίσεις της εσωτερικής αγοράς. Αυτό ισχύει και για τα προϊόντα που εισέρχονται αλλά και για τα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό αυτής της ε, εσωτερικής αγοράς υπάρχει ένα κομμάτι θα έλεγα της οικονομικής δραστηριότητας που εξαρτάται από τις δημόσιες προμήθειες. Πράγματι πιστεύω ότι ο σεβασμός των κανόνων στον τομέα των δημοσίων προμηθειών και η πρόοδος την οποία μπορούμε να σημειώσουμε στα πλαίσια της των ηλεκτρονικών διοργανώσεων αυτών των προμηθειών είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Πριν μερικές μέρες είχατε έρθει ορισμένοι από εσά στο workshop που κάναμε σε συνεργασία με τον Ετσεβερία και τον Ταραμπελά και πράγματι είχαμε συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι αν μπορέσουμε από κοινού επί τη βάση των κειμένων μας να συστηματοποιήσουμε και να αναπτύξουμε με γενικό τρόπο την ηλεκτρονική, τις ηλεκτρονικές διαδικασίες των δημοσίων προμηθειών, μπορούμε να εξοικονομήσουμε με όλες τις τοπικές και περιφερειακές αρχές μέσω αυτής της ψηφιοποίησης και γενίκευσης των διαδικασιών 100 δις κατέτος λέει ο Λοιπόν, συμφωνώ και με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σβάμπ για τους στόχους της εσωτερικής αγοράς και για το πόσο θα είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό προσπαθούμε στα πλαίσια όλων των διαδικασιών μας να ακαλύψουμε τις ανάγκες και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις δυνατότητες επενδύσεων στις επιχειρήσεις αυτές. Να πω στον κύριο Γκούσταυσον ότι η ενιαία αγορά τι ακριβώς είναι. Είναι αν θέλετε η πλατφόρμα, είναι ακριβώς τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομούμε τις επιμέρους πολιτικές. Έχει σημασία το πάτωμα πάνω στο οποίο πατάμε να είναι σταθερό, να είναι συμπαγές. Έτσι μόνο θα είναι αποτελεσματική οικονομική μας δραστηριότητα. Και έτσι ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε και για την λεγόμενη πράσινη πολιτική στην οποία αναφέρθηκε ο Γκούσταυσον στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Εδώ έχω και το εγχειρίδιο για τους 12 μοχλούς αυτής της ενιαίας πράξης για την εσωτερική αγορά εγώ εδώ έχουμε συμπεριλάβει ακριβώς τα θεμέλια μιας κοινωνικής ανταγωνιστικής οικονομίας της αγοράς. Επιμένουμε σε αυτές τις λέξεις που προανέφερα. Λοιπόν, θα δείτε ακριβώς αυτούς τους 12 μοχλούς που θεωρούμε ε, χρήσιμους στα πλαίσια ε, του συμφώνου αυτού ε, υπαρίθμου 2. Να πω λοιπόν κύριε Γκάλπες ότι είναι αποτελεσματική πράγματι η έκθεση Μπουσούτιλ όπως ακριβώς το εξέφρασε και ο κύριος Σβάμπ. Πρέπει κάθε φορά να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται και κάνουμε αυτή την προσπάθεια του screening εκ των προτέρων ελέγχου έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις δυνατότητες εφαρμογής της οδηγίας και στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στον τομέα της εσωτερικής αγοράς και γι' αυτό με την κυρία Σάλντε Μόζε προετοιμαζόμαστε για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο Συμβούλιο επαναλαμβάνω παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σαν συνομοθέτης. Επαναλαμβάνω, Επιτροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο πρέπει να δράσουμε αποτελεσματικά επί τη βάση των 40 εγγράφων κειμένων που είναι σε αυτήν εδώ την προσούρα, σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο που όλοι έχουμε εδώ και μήνες μπροστά μας. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο ε, καταργώντας ε, τα εμπόδια που είπε, στα οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος Χάρμπορ, γιατί τα εμπόδια αυτά είναι χαμένες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, χαμένες ευκαιρίες για την απασχόληση και στους δύσκολους αυτούς καιρούς δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε ευκαιρίες. Όπως είπε ο κύριος Μπουσούτη λοιπόν, πρέπει μαζί με τα κράτη-μέλη να θέσουμε σε εφαρμογή όλα τα κείμενα που αφορούν και έχουν ψηφιστεί ε, την εσωτερική αγορά και να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο τομέα προς τομέα, δραστηριότητα προς δραστηριότητα, αναδραστηριότητα, έτσι ώστε η εσωτερική αυτή αγορά να γίνει πιο αποτελεσματική. Νομίζω κυρίες και κύριοι ότι εκεί ακριβώς έχουμε την πιο απτή και την πιο θα έλεγα ε, κοντινή μας δυνατότητα για ανάπτυξη. Λόγο στον μας, τον κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέσσερα λεπτά. Μου δώσατε έτσι μου είπα. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Θα αρχίσω κύριε Πρόεδρε με ευχαριστίες προς τον Επίτροπο Μπαρνιέ και προς όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έλαβαν τον λόγο σε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση, όλους εκείνους οι οποίοι χωρίς σχεδόν καμία επιφύλαξη είπαν ότι είναι υπέρ, αλλά ευχαριστώ και εκείνους που έχουν κάποιες επιφυλάξεις, θα κατεβάσουν και κάποιες ε, α, επιτροπολογίε και θα επανέλθουμε σε αυτά. Οπότε πρώτα πρώτα για να επανέλθουμε ή σε αυτό το παράδειγμα το οποίο επεσήμανε ο, ο κ. Μπαρνία σε σχέση με αυτή τη συζήτηση που είπε ότι έχουμε εδώ ένα παράδοξο το οποίο από τη μια μεριά είναι ένα παράδοξο και όλοι καταλαβαίνουμε τις δυνατότητες της νέας αγοράς, κάτι το οποίο σχεδόν όλοι το ξέρουμε. Όμως από την άλλη μεριά γνωρίζουμε ότι η εσωτερική αγορά πολλές φορές είναι το πρώτο θύμα στην περίπτωση που τα πράγματα πάνε στραβά. Το πρώτο θύμα κάποιων ε, τάσεων προστατευτισμού. Να ένα παράδοξο που θα πρέπει να το επιλύσουμε, ένας φραγμός τον οποίο θα πρέπει να άρουμε. Πάντως έχουμε τρεις τρόπους κατά τη γνώμη που μπορούμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Πρώτα-πρώτα την μεταφορά της νομοθεσίας θα πρέπει να ε, γίνεται έγκαιρη η μεταφορά της κοινωνικής νομοθεσίας στην εσωτερική τάξη. γιατί αν δεν γίνει αυτό τότε υπάρχει πρόβλημα. Κατά δεύτερο λόγο, θα πρέπει να ε, εφαρμόζονται σωστά, αποτελεσματικά τα νομοθετήματα. Ιδάλλως δεν έχει νόημα να θεσπίζονται Αυτή η νομικά τα τρίτο λόγο επίσης θα πρέπει και επιχείρηση αλλά και οι Ευρωπαίοι να έχουν τα μέτρα προς άσκηση κάποιου ενδίκου μέσου όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Κάποιοι συνάδελφοι επίση διατύπωσαν κάποιε επιλύσει όσον αφορά την τροπολογία η οποία πρόκειται να ε, υποβληθεί και για να δούμε, για να διασκεδάσω του εμβολίου του, διότι ε, έχει τα εξή και λέει ότι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα πρέπει να συγκροτήσει μια διαδικασία επί παραβάση συνοπτική και θα πρέπει επίση και, και τονίζεται θα πρέπει να, να, να, να μελετήσει την συγκρότηση επίση ε, μια ε, μονάδα, μια υπηρεσία, ώστε να διώκονται οι πράξεις παραβίαση και παραπομπήσεις στο δικαστήριο όταν συμφωνεί το σώμα του Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόκειται για μια τροπολογία η οποία ε, έρχεται να συμπληρώσει την ε, διαδικασία θέσπισης ε, της συνοπτικής διαδικασίας η παραβάση θα πρέπει να την κοιτάξουμε τη διαδικασία διότι έτσι θα απελευθερώσουμε την Επιτροπή από την πολιτική πίεση πάρα πολύ συχνά αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν πρέπει να κάνει μια καλύτερη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο, όταν πρέπει να κάνει κάποιες διαπραγματεύσεις για αυτή τη διαδικασία των ε, ε, επιπαραβιάσει και πολλές φορές ε, βραδύνει πάρα πολύ ολοκλήρωση τη διαδικασία αυτή. Οπότε δεν πρόκειται, όπω είπε η κυρία Ράπτη, περί διαδικασία υποβολή κυρώσεων. Πρόκειται περί αποπολιτικοποίηση αυτή τη διαδικασία, περί, περί του πώ θα την καταστήσουμε πιο διεκπαιρεωτική, πιο γρήγορη δεν είναι μια απειλή, είναι απλώ μια βοήθεια να γίνει πιο καλή η ιστορική αγορά και γιατί είπαμε να γίνει αυτό εδώ και τώρα, διότι αν δεν κάνουμε κάτι εδώ και τώρα, τότε, τότε, τότε το παιχνίδι θα χαθεί και είναι κατακλείδη, θα πρέπει να συμφωνήσω προς όλους του αδελφούς οι οποίοι είπαν ότι το βασικό ατού τη Ευρώπη είναι η εσωτερική αγορά. Το δε πρόβλημα που έχουμε το αντιμετωπίσουμε είναι το να εξασφαλίσουμε ότι η εσωτερική αγορά θα είναι λειτουργική για όλους. Άρα να δράξουμε αυτή την ευκαιρία. Μια που τρέχουμε την 20η επέτειο και έτσι να μπορέσουμε να εξεύρουμε την πολιτική βούληση έτσι οι τελευταία ψεγάδια, τελευταία μειονεκτήματα να αρθούν και έτσι να γίνει μια αυθεντικά ενή αγορά η οποία να μπορεί να μας οδηγεί στον δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας που όλοι προσδοκούμε. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση γύρω από την έκθεση του κυρίου Μπουσουτήλ για τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς ολοκληρώθηκε και θέλω να σας ενημερώσω ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και περνάμε στο επόμενο σημείο